να συγχαρώ την εισηγήτρια που ε, εξακολουθεί να υπάρχει για το δικαίωμα της απεργίας. Εν συντομία, θεωρώ ότι είναι ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός, που είναι όμως πολύ σημαντικό για τον τομέα αυτόν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για την ομιλία σας αυτά, αυτή. Τρεμόζα Μπαρτσέλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.